για του ενιαίου κανόνε και την ενιαία διαδικασία επιστοτικών ιδρυμάτων και ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων στο πλαίσιο ενό ενιαίου μηχανισμού εξυγίανση και ενό ενιαίου ταμείου εξυγίανση τραπεζών. Πρόκειται για το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων. Κυρίε και κύριοι, θα ήθελα να σα επισημάνω ότι δεν προβλέπεται διαδικασία καρστιάη κατά το σημείο αυτό τη συζήτηση, ούτε η διαδικασία τη πλε κάρτας. Δεν εφαρμόζεται. Δεν ξέρω γιατί, αλλά πάντως αυτό έχει αποφασιστεί. Οι ομιλητέ τώρα εκ μέρου των ομάδων. Κυρία Βόρτμαν Κόλ, εκ μέρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο. Σα Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θεωρούμε ότι είναι επίγουσα η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης και μάλιστα πριν τις ευρωεκλογέ. Γι' αυτό και σήμερα θα πρέπει να επιβεβαιώσουμε και να διατρανώσουμε την ισχυρή διαπραγματευτική μας εντολή για τις διαπραγματεύσεις για τον ενιαίο μηχανισμό εποπτείας, ε, μηχανισμό εξυγίανσης. Ούτως ή άλλως οι αρμόδιες επιτροπές υπερψήφισαν με μεγάλη πλειοψηφία αυτή τη διαπραγματευτική εντολή. Στη σημερινή ψηφοφορία θα πρέπει να κρούσουμε τον κόδωνα του κινδύνου στο Συμβούλιο και να το αφυπνίσουμε. Άλλωστε η συζήτηση της Τρίτης επιβεβαίωσε αυτή τη ε, μεγάλη συνένεση. Και ο αντιπρόεδρος της ελληνικής κυβέρνησης ε, δυστυχώς ε, ήταν, μάλιστα, συγγνώμη, ήταν παρόν στην συζήτηση, κάτι που δείχνει τι μεγάλη προτεραιότητα έχει για την ελληνική Προεδρία ο σχετικό κανονισμό. Και μάλιστα το Συμβούλιο, η Προεδρία μα είπε ότι είναι πρόθυμη να εργαστεί επικοδομητικά μαζί μα για μια συμφωνία. Αλλά η ελληνική Προεδρία δεν δύναται να κάνει τις διαπραγματεύσεις χωρίς σημαντική εντολή από το Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ. Αλλά υπάρχει η αίσθηση του κατεπήγοντος, γιατί οι αγορές μας παρακολουθούν. Όταν, ε, όταν είχαμε το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, διορθώσαμε κάποιες διαρθρωτικές αδυναμίες και περάσαμε σε κοινού εποπτικού κανόνε, αφαιρώντα την εποπτεία της τι εξασφαλίζοντα μεγαλύτερη αντικειμενικότητα και σε τελική ανάλυση συμφωνήσαμε ότι χάρη στι διατάξει αυτέ κάναμε το εξάπτυχο μια καλή συμφωνία. Τώρα το Συμβούλιο προτείνει το αντίθετο. Να αφήσουμε τι κρίσιμε αποφάσει για την εξυγίαση προβληματικών τραπεζών στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών. Πολύ αμφιβάλλω όμω αν μια τέτοια λύση θα μας οδηγήσει σε μια αποτελεσματική και αντικειμενική διαδικασία λήψης αποφάσεων. Και πώς θα λειτουργήσει κάτι τέτοιο όταν μια τράπεζα πρέπει να καθαριστεί μέσα σε δύο μέρες, 48 ώρες. Μία τέτοια πρόταση θα μπορούσε να υπονομεύσει την αποτελεσματική εφαρμογή των μηχανισμών εξυγίανση. Θέλουμε να μπορέσει να εφαρμοστεί το bail-in, η ώστε να πληρώνουν οι μέτοχοι και οι επενδυτές, αλλά να εφαρμόζεται το ίδιο ο μηχανισμός αυτός στις προβληματικές τράπεζες, άσχετα με το κράτος μέλος το οποίο δραστηριοποιούνται. Η μεταχείριση θα πρέπει να ισχύει όπου χρειάζεται και στην πρόσβαση στο Ταμείο Εξυγένσης. Και εκεί η θέση του Συμβουλίου υστερεί σε σχέση με τη δική μα. γιατί το Ταμείο έχει ε, κατακαιρματιστεί άκαμπτα σε εθνικά τμήματα. Έτσι θα ενισχυθεί ο κακός ε, σύνδεσμος μεταξύ δημόσιου χρέους και τραπεζών να διαρριχθεί. Άλλωστε, η Υπάρχει κίνδυνο ε, και για τη φήμη τη νέα ε, αρχή εξυγίαση. Δεν θέλουμε ήδη να υπονομευθεί η τράπεζα πριν λειτουργήσει. Το ενιαίο ταμείο θα πρέπει να αρχίσει να λειτουργεί από την έναρξη λειτουργία και του ενιαίου μηχανισμού εξυγίαση ε, με κοινή ανάθεση των εισφορών των τραπεζών, αντί να έχουμε δεκαετή εθνική ανάληψη. Και φυσικά χρειάζεται και μια δανειοδοτική διευκόλυνση. Η Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή ψήφισε σαφέστατα υπέρ ενός ενιαίου μηχανισμού εξυγίανσης. Με ένα ενιαίο ταμείο εξυγίανσης, όπου μια τράπεζα θα μπορεί να καθαρίζεται και μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο. Ένα σύστημα που θα πληρώνουν οι ίδιες οι τράπεζες θα χρηματοδοτούν τη διαδικασία αυτή. Και η ομάδα μα θέλει να προστατεύσει τους φορολογούμενου, να μην πληρώνουν αυτοί τα σπασμένα των προβληματικών τραπεζών. Το Συμβούλιο ε, εισήγαγε μια προσωρινή διακυβερνητική συμφωνία. Προσωρινή μεν, αλλά παρόλα αυτά είμαστε πολύ επιφυλακτικοί απέναντι στη συμφωνία αυτή, γιατί εμείς δεν πιστεύουμε σε διακυβερνητικές λύσεις. Εκτός κι αν μας πείσει κάποιος ότι είναι απολύτως απαραίτητη μια τέτοια λύση για να εκπληρωθούν κάποιες συνταγματικές ανάγκες και φυσικά εφόσον έχουμε πιστεί για τον νομότυπο μιας τέτοιας λύσης. Έχω κάποια κατανόηση για κάποιες συνταγματικές επιφυλάξεις ορισμένων κρατών μελών ό,τι αφορά την ε, μεταφορά των συνεισφορών από τις τράπεζες στο Ευρωπαϊκό Ταμείο. Αλλά δεν μπορούμε να δεχτούμε μια διακυβερνητική συμφωνία που αφαιρεί πολύ σημαντικά και κρίσιμα στοιχεία του ενιαίου μηχανισμού εξυγίανσης από το, ταμείο, από το μηχανισμό αυτό και το μεταφέρει στα κράτη-μέλη. Η διαπραγματευτική τράπεζα βρίσκεται εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όχι στο κτίριο του Συμβουλίου. Οι τριμερεί διάλογοι με την Ελληνική Προεδρία είναι το κατάλληλο φόρουμ διαπραγμάτευση, κατά τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και θα ήθελα να καλωσορίσω την επικοδομητική στάση του Επιτρόπου Μπαρνιέ στη συζήτηση τη Τρίτη. γιατί η δική σα αρχική πρόταση για ενιαίο μηχανισμό εξυγίαση είναι η σωστή βάση και δείχνει το σωστό δρόμο. Και μάλιστα έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στην επιμονή σας για ένα αξιόπιστο και αποτελεσματικό σύστημα. Και πιστεύουμε ότι εστερνίζεστε τη γνώμη μας ότι μια συμφωνία είναι κατεπίγουσα και θα πρέπει να ληφθεί κατεπηγόντως, αλλά όχι πάση θυσία. Η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης είναι ύψιστη προτεραιότητα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος λίγους μήνες πριν από τις ευρωεκλογές. Ο ενιαίος μηχανισμός εξυγένσης είναι το τελευταίο δομικό κομμάτι αυτή τη συμφωνία. Θα πρέπει να θεσπιστεί για να εξασφαλίσουμε την αξιοπιστία και ένα ασφαλέ χρηματοπιστωτικό σύστημα με καλύτερη πρόσβαση των ε, νοικοκυριών και των επιχειρήσεών μα στο δανεισμό. Θέλουμε επίση να προστατεύσουμε του συμπολίτε μα και τι καταθέσει του από χρεοκοπημένε προβληματικέ τράπεζε. Θα πρέπει με την Τραπεζική Ένωση να επιταχύνουμε την οικονομική ανάπτυξη και να αποκαταστήσουμε την ε, εμπιστοσύνη. Είμαστε έχουμε συνείδηση της μεγάλης ευθύνης που μας ε, βαρύνει. Έχουμε μια συμφωνία, θα ψηφίσουμε τώρα αυτή τη συμφωνία για να δώσουμε ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας. Η γραμμή μας που συμφωνήθηκε στην Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή ευελπιστούμε ότι θα τύχει πλήρους υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμείς δεν τροποποιούμε τη διαπραγματευτική μας εντολή, επαναλαμβάνουμε τις απόψεις μας όπως ε, τις παρουσίες οικιακών πέρυσι το Δεκέμβριο. Δεν ολοκληρώνουμε την πρώτη ανάγνωση, κρατούμε την πόρτα ανοιχτή. Και επαναλαμβάνω, θα πρέπει να αφυπνιστεί το Συμβούλιο. Το Κοινοβούλιο είναι ανοιχτό και έτοιμο για επιτάχυση των διαπραγματεύσεων και ε, σύναψη συμφωνίε πριν τι ευρωεκλογέ. Θα, είμαστε, θα δείξουμε πυγμή αποφασιστικότητα, αλλά θα είμαστε και επικοδομητικοί. Δεν μπορούμε όμω να δεχθούμε οποιαδήποτε συμφωνία. Η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Τράπεζας μας ενδιαφέρει, αλλά θα πρέπει να γίνει με σωστό τρόπο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Βορτμαν Κόλ. Και τώρα το λόγο εκ μέρου τη ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, κύριο Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Πίτροπε. Το μήνυμα μας είναι σαφέστατο, την πολιτική μας ομάδα, Θέλουμε καταρχάς μια λύση. Αλλά όχι αυτή που προτείνει το Συμβούλιο. Δεν είναι αποδεκτή η λύση του Συμβουλίου. Δεύτερον, θέλουμε μια λύση για την εντολή από το Συμβούλιο. Και αν θέλει στα σοβαρά να λυθεί το θέμα το Συμβούλιο, πρέπει ταχύτατα να δώσει εντολή για διαπραγμάτευση στην Ελληνική Προεδρία. Εάν στραφούμε στην εποχή όπου αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ότι θέλει την Τραπεζική Ένωση και αναλογιστούμε πόσοι μήνες έχουν περάσει μέχρι τώρα, προφανώς δεν είναι δική μας ευθύνη, δεν είναι δικό μας το σφάλμα που δεν υπάρχει ακόμη Τραπεζική Ένωση. Αυτό οφείλεται στο... Κύριε Σφόπο, το διακόπτει ο Πρόεδρος. Με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά έχουμε ένα τεχνικό ζήτημα. Έχουν εμπερδευτεί τα κανάλια των, ε, της γαλλικής και της γερμανικής γλώσσας. ο τεχνικός μπορεί να κάνει μια προσπάθεια. Ο κύριος Λάγκεν διαμαρτύρεται γιατί δεν σας ακούει. Ακούει γαλλικά αντί για γερμανικά. Ο κύριος Λάγκεν χωρίς μικρόφωνο. Αυτό είναι το πρόβλημα που δεν έχουμε εδώ παρόν το Συμβούλιο. Αυτό είναι το κύριο πρόβλημα. Τώρα τι σχέση έχει αυτό με την, με την παρουσία του Συμβουλίου λέει ο πρόεδρος. Μα, το είχατε κάπως επισημάνει στην αρχή της παρέμβασης. Εγώ προσπάθησα να σας βοηθήσω για να δούμε τι γίνεται το μεταξύ με, την, με τα κανάλια της Δερμηνίας. Ο κύριος Λάγκεν είναι ικανοποιημένος. Πολύ ωραία λέει και ο κύριος Βόμποντα. Συνεχίζω. Ποιο είναι λοιπόν το πραγματικό πρόβλημα. Το πραγματικό πρόβλημα είναι το εξή για μας. Το Συμβούλιο δεν θέλει το πραγματικά ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο, το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρουν περισσότερες εξουσίες στο θέμα αυτό. Και είναι κρίμα αυτό και παράδοξο, διότι είναι ευρωπαϊκό το θέμα. Όλο και πιο συχνά λοιπόν στο Συμβούλιο οι Υπουργοί λένε ναι, επί τη ουσία μπορεί να συμφωνούμε, αλλά θα το αναλάβουμε εμεί. Εμεί που είμαστε Υπουργοί. Αλλά θα πρέπει να εξηγήσουν στου πολίτε και εδώ, στου παρισταμένου επισκέπτε, στα θεωρία, γιατί δεν είναι αποτελεσματικέ οι αποφάσει του. Διότι για να καταλήξουν σε μια συμφωνία στο Συμβούλιο, παρότι είναι μόλι 28, δυσκολεύονται πολύ περισσότερο από ότι εμεί εδώ στο Κοινοβούλιο με σαφεί ψηφοφορίε και καλή συνεργασία μεταξύ μα. Οι προτάσει λοιπόν του Συμφωνιού δεν είναι αποτελεσματικέ και γι' αυτό και απορρίπτονται. Επέλεξε ω νομική βάση το Συμβούλιο ένα άρθρο που μπορεί να είναι ε, ε ορθή νομική βάση, αλλά πολιτικά επιλεγμένη μια άλλη νομική βάση που θα εξασφάλιζε την κοινοτική μέθοδο, δηλαδή με κυρίαρχο ρόλο για την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο, επίση θα λειτουργούσε πολύ καλά. Γιατί λοιπόν επέλεξαν τη νομική βάση τη διακυβερνητική συνεργασία, γιατί θέλουν να διατηρήσουν την επιρροή του. Πλην όμω το, το ευρωπαϊκό ε, τραπεζικό σύστημα δεν είναι πια στα χέρια των κρατών μελών. Δεν είναι εθνικό τραπεζικό σύστημα, είναι ευρωπαϊκό και γι' αυτό δεν μπορεί να βρει λύσει σε εθνικά χέρια. Επίση, θα πρέπει να εξηγήσουμε στους πολίτες μας το εξή ότι η Τραπεζική Ένωση δεν έχει στόχο να εξυπηρετήσει τις τράπεζες, αλλά να προστατεύσει του πολίτες, τους πολίτες που φοβούνται ότι θα χάσουν τις καταθέσεις τους, τους πολίτες που φοβούνται ότι δεν θα μπορούν να πάρουν ένα δάνειο και ότι θα έχουν δυσκολίες όταν αποτυγχάνουν οι τράπεζες να διαδραματίσουν το ρόλο τους. Αυτό λοιπόν έχουμε λησμονήσει να πούμε στους πολίτες ότι η Τραπεζική Ένωση έχει στόχο να εξυπηρετήσει τον πολίτη και όχι την τράπεζα. Και γιατί χρειάζεται μια ισχυρή και ευρωπαϊκή λύση. Το βλέπουμε και πάλι από τους Financial Times ε, που διαβάζω και που δείχνουν ε, μια κατάσταση από το Ηνωμένο Βασίλειο, αγαπητέ κύριε κάλα, ότι κάποιοι προσπαθούν να αντιπαρέλθουν ρυθμίσεις που έχουν περάσει για τα μπόνους, επί παραδείγματι, των μάνατζερ ε, των μεγάλων επιχειρήσεων που περιορίζονται και προσπαθούν με άλλους τρόπους νομότυπους, νόμιμους τυπικά, αλλά πάντως όχι σωστούς, να αντιπαρέλθουν την νομοθεσία. Ε, αυτό λοιπόν πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τώρα είναι η ώρα, όπως υπόθηκε, να βρούμε λύση η οποία δεν θα επιβαρύνει τον φορολογούμενο, αλλά τις τράπεζες της ίδιας. Και όπως είπα, δεν είναι καλός ο μηχανισμός. Θα χρειάζεται μια μακρά διαδικασία πριν ε, καταλήξουμε σε λύση, άρα θα πρέπει να βελτιώσουμε τον μηχανισμό. Εμείς με χαρά είδαμε τη διάταξη που έλεγε ότι θα μπορούσε η Επιτροπή να αποφασίσει αν χρειάζεται η ακαθάριση μια τράπεζας. Πρέπει να επανέλθει λοιπόν αυτή η διάταξη. Και ή μη τι άλλο να βρεθεί μια διαφορετική λύση από αυτή που έχουμε τώρα, γιατί είναι υπερβολικά περίπλοκη. Α φανταστούμε ότι ξεσπάει σε μια πόλη πυρκαγιά και θα πρέπει να συγκληθεί το Δημοτικό Συμβούλιο για να αποφασίσει αν θα πρέπει να ληφθεί μέτρο. Έμα ε, όταν έχουμε μια κατάσταση, σε ένα νοσοκομείο, όπω είπε και ο πρόεδρο νωρίτερα, δεν πάμε να καλέσουμε το διοικητικό συμβούλιο του νοσοκομείου να, κάνει, να λάβει αποφάσει για το τι θα πρέπει να κάνει για το συγκεκριμένο ασθενή. Ο γιατρό που τον έχει στα χέρια του θα αποφασίσει πώ θα χειριστεί την κέρια εκείνη στιγμή την κατάσταση. Επίση το χρονοδιάγραμμα. Τα 10 χρόνια παρά είναι μακροδιάστημα για να συσταθεί αυτό το ταμείο που ούτω ή άλλω δεν θα είναι επαρκέ. Και η δυνατότητα για περιορισμό στα 5 χρόνια τη περίοδου για τη σύσταση που μα λένε κάποιοι θα σημαίνει ότι κάποιες τράπεζες στα πιο ασθενή κράτη θα πρέπει να καταβάλουν πολύ μεγαλύτερες εισφορές. Ωραία, ωραία. Ας βάλουμε λοιπόν ένα όριο. Ένα όριο βιώσιμο για τις τράπεζες στη συμμετοχή τους, στην δυνατότητα το Ταμείο να στήσει εισφορές και στη δυνατότητα του Ταμείου να αντιδράσει στις παριστάμενες ανάγκες. Αυτό νομίζω ότι είναι μια ορθολογική λύση. με τον μηχανισμό προστασίας νομίζω ότι δίνουμε τη λύση. Και θα ήθελα επίσης να πω ότι υπάρχει ενότητα και στεναρές, σαφείς θέσεις. Δεν συμφωνείτε! Σαφείς θέσεις από πλευράς διαπραγματευτική ομάδας και αυτό είναι το κύριο πλεονέκτημα που έχει το Κοινοβουλίο να παρουσιάσει. Η διαπραγματευτική μας ομάδα πρέπει να έχει σαφή θέση και αυτή είναι η θέση τη πολιτική μα ομάδα είναι καλύτερη η μη λύση από μια κακή λύση. Δεν είμαστε διατεθειμένοι πάση θυσία να δεχθούμε κάποια λύση, ακόμη και αν αυτή είναι κακή. Μόνο και μόνο για να την εξασφαλίσουμε γρήγορα. Θα ήταν πολύ καλύτερο να καθυστερήσουμε για να έχουμε μια καλή λύση αργότερα. Αυτή είναι η θέση τη ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ζητούμε από το Συμβούλιο να δώσει ταχύτατα εντολή και καλούμε το Συμβούλιο να μην περιμένει μέχρι τη 17η-18η Φεβρουαρίου για την εντολή. Α ξεκινήσει από την επόμενη εβδομάδα για να ξεκινήσουμε και εμεί τι διαπραγματεύσει. Όπω είπα, θέλουμε λύση, δεν δεχόμαστε όμω και δεν είμαστε διατεθειμένοι να δεχθούμε μια λύση κακή γιατί η ανυπαρξία λύση, η μη επίλυση είναι για μας καλύτερη από μια κακή λύση. Ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους των φιλελευθέρων και δημοκρατών ο κύριος Φερχόφστατ έχει το λόγο. Πρόεδρε, το πρώτο θέμα θέλω να θίξω και να ρωτήσω είναι πού είναι το Συμβούλιο. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Εδώ στέλνουμε ένα μήνυμα. Δεν είναι μήνυμα για τον κύριο Μπαρνιέ, διότι ο κύριο Μπαρνιέ είναι 100% πίσω μα, το στηρίζει και έχουμε ίδιε απόψει Έχουμε ένα μήνυμα για ποιον, για το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο γιατί απουσιάζει. Ε, δεν είναι για τα μέσα ενημέρωση, κύριε Κάρα. Ίσως εσεί θα το κάνετε για τα μέσα ενημέρωση. Έτσι είστε κατά τη τραπεζική ενώσεω. Άρα το ότι απουσιάζει η Προεδρία. Πρέπει να μα κάνει νέα πρόταση η Προεδρία. Και ο κύριο Σβόμποντα έχει απόλυτα δίκιο. Είναι απαράδεκτο ότι θα χρειαστούμε τώρα μέχρι πότε, πότε έχουμε το νέο ΕΚΟΦΗΝ κύριε Μπαρνιέ, 17 17 Φεβρουαρίου πριν να δοθεί η νέα εντολή. 14 μέρες χαμένες. Ξανά. Πάνω από τους μήνες που χάσαμε. Διότι αποφάσισε το Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2012. Το Συμβούλιο Τραπεζική Ένωση. Ιούνιο 2012. Και σήμερα δεν είμαστε σε θέση να δώσουμε ε, να δοθεί νέα εντολή για να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσει του Κοινοβούλιο. Για να είμαστε ειλικρινεί, Ήδη είπαμε επανειλημμένω ότι η πρόταση του Συμβουλίου δεν ήταν αποδεκτή και χρειαζόταν μια άλλη. Και ποιο είναι το δραματικό σημείο. Ότι εδώ και έξι χρόνια, έξι χρόνια ξεκίνησε η χρηματοδοτική κρίση. Εδώ και έξι χρόνια. Και ακόμα δεν έχουμε μια λύση για την τραπεζική κρίση. Οι Αμερικανοί αμέσω κινήθηκαν. Το πρώτο που έκαναν οι Αμερικανοί εντό ενό έτου μετά την έναρξη τη κρίσης ήταν να κεφαλοποιήσουν τι τράπεζε και να λύσουν το πρόβλημα. Το έκαναν και οι Σουηδοί μετά από τη δική του κρίση στο τραπεζικό τομέα και το στεγαστικό. Στα στεγαστικά δάνεια. Και εμεί ε, ακολουθούμε του Ιάπωνε. Περίμενα 15 χρόνια μέχρι να ανακεφαλοποιήσουν τι ε, ε τράπεζε. Αποτελμάτωση οικονομική ήταν το αποτέλεσμα αυτή τη προσέγγιση. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, εν ονόματι του Κοινοβουλίου, του Ενωμένου Κοινοβουλίου, πραγματικά σας ζητώ να στείλετε μία επιστολή προς την Προεδρία του Συμβουλίου και να πείτε, προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και να πείτε ότι είναι αυτό απαράδεκτο και ζητούμε από το Συμβούλιο να επιταχύνουν τις διαπραγματεύσεις εντός του Συμβουλίου ώστε να μας ε, δοθεί μια νέα εντολή. Λοιπόν, μετά... Ε, ε, λοιπόν, το χρονοδιάγραμμα η ταχύτητα είναι σαν τράμπαν η ταχύτητα της προτάσεως του ε, Συμβουλίου. Πολύ ε, αργοκίνητη διαδικασία σαν τράμπαντ. Χρειάζεσαι Μακλάρεν ή Φεράρι να κινηθείς για να λύσεις τα προβλήματα. Και να τα λύσεις ένα Σαββατοκύριακο. Και μετά όσον αφορά τη νομική βάση, νομίζω ότι υπάρχει μόνο μια καλή νομική βάση, το 114, γιατί διότι τα ποσά είναι, οφείλονται σε ιδιωτικές συνεισφορές, δεν είναι των τραπεζών. Ε, δεν θέλουμε να χρησιμοποιηθούν λοιπόν δημόσιοι πόροι. Άρθρο 114, 114 είναι η σωστή νομική βάση. Άκουσα ήδη να λέγεται ότι κάποιοι συμφωνούν στο μεν, συμβιβάζονται στο άλλο, ίσως να έχουμε μια ρήτα σταδιακής εξάλληψης, ούτως ώστε να εμπέσει σε κοινοτικό δίκαιο αργότερα η νομοθεσία. Λέμε, ξεκινάμε αυτό το σύστημα, έχει ξαναγίνει αυτό, αλλά σε 2, 4, 5 χρόνια θα πρέπει το σύστημα να ε, καταλήξει σε κοινοτικό δίκαιο. Σε αυτό να είναι το αποτέλεσμα. Είναι καλό. Δεν ξέρω. Ίσως είναι καλύτερα από άλλες λύσεις. Α ξεκινήσουν διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο και να μείνουμε στο άρθρο 114, νομική υπηρεσία του Συμβουλίου μαζί με την νομική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την νομική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αν και οι τρεις νομικές υπηρεσίες λένε το ίδιο πράγμα, είναι θαύμα θα έλεγα αυτό. Διότι κανονικά οι νομικές υπηρεσίες πάντα έχουν διαφορετικέ απόψεις. Αυτή τη φορά έχουν την ίδια άποψη. Και μόνο επειδή μια χώρα ε, ε, ε, είναι αντίθετη εξετάζουμε ξανά το ενδεχόμενο διακυβερνητικού συστήματος εκτός των συνθήκων. Και αυτό έχει αρνητική επιρροή όσον αφορά τις εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. ο κύριος Κονβέντιτ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, Δίκαιο έχει ο Γκίφερ Χόφστατ από τον Ιούνιο του 2012. Και ξέρετε γιατί δράει έτσι το Συμβούλιο. Γιατί ξέρει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Συμβούλιο γνωρίζει ότι αν πιέσει το ε, Κοινοβούλιο στα, όρια του και το οθεί στα όρια του, γιατί είπε δεν θα απορρίψετε την Τραπεζική Ένωση. Έτσι είχε γίνει και με τον προπολογισμό. Έχω άπειρα παραδείγματα. Και την τελευταία στιγμή θα δείτε πώς ε, θα υιοθετηθεί η μισή τουλάχιστον πρόταση του Συμβουλίου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενδεχομένω με αυτά που είπε ο Γκί. Λέγοντα θα δούμε σε 3, 10, 50 χρόνια, δεν ξέρω κι εγώ πότε, θα δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Γι' αυτό δεν σπέβδει το Συμβούλιο, γι' αυτό δεν βιάζεται, γιατί όσο πλησιάζουμε προ τι εκλογέ και εκπνέει η κοινοβουλευτική μα θητεία, ξέρει το Συμβούλιο ότι θα κερδίσει, θα περάσει δική του θέση. Επίσης γνωρίζουμε ότι έχουμε 294, ε, 114, είναι περίπλοκες οι διαδικασίες. Το θέμα δεν, δεν πρόκειται για δημόσια χρήματα. Για, ας μην μας ε, ε, ενοχλεί η, Γερμανία. Δεν έχει καμία σχέση εκεί το Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο. Πρόκειται για ιδιωτικά κονδύλια, για πολυεθνικές εταιρείες. Ξέρω, η Deutsche Bank, λέγεται βέβαια Deutsche Bank Γερμανική Τράπεζα, αλλά έχει δραστηριότητε παντού στην Ευρώπη. Η Unicredit έχει το μεγαλύτερο τζίρο, το μεγαλύτερο κύκλο εργασιών στη Γερμανία. Ας α, μην μας παραμυθιάζουν λοιπόν που με το ότι θέλουν να προστατεύσουν τα ε, χρήματα των φορολογουμένων. Όχι, θέλουν να βρουν ένα, έναν ε, μηχανισμό εκαθάρισης, θέλουμε να βρούμε μηχανισμό εκαθάρισης για τις ιδιωτικέ τράπεζες. Γι' αυτό και οι χώρες δεν θα πρέπει να βάζουν σημαία στο, την εθνική του σημαία σε αυτό το μηχανισμό. Επίσης το, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να είναι σαφές. Θέλουμε να οργανώσουμε την προστασία των πολιτών και να οργανώσουμε το σύστημα ώστε οι τράπεζες να μην χρησιμοποιούν τα κονδύλια των φορολογουμένων, να μην στρέφονται τις χώρες και να λένε βρισκόμαστε στα πρόθυρα χρεοκοπίας, σώστε μας. Χρειαζόμαστε έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό. Και αυτό είναι το περίεργο. Αν όπω πρότειναν μερικέ χώρε στο Συμβούλιο, το κάνουμε ένα χώρα, το κατακαιρματίσουμε το σύστημα, θα δείξουμε και πάλι την ανικανότητά μας να δείξουμε αλληλεγγύη. Οι πιο αδύναμοι θα παραμείνουν αδύνατοι και οι ισχυρότεροι θα παραμείνουν ισχυροί. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε με αυτό που κάνουμε. Ε, όχι, αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να το απορρίψει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο μόνος τρόπος για να κερδίσουμε είναι να πούμε και να επαναλάβουμε και να διατρανώσουμε ότι προτιμούμε καθόλου λύση από μια κακή λύση. Αν καταφέρουμε να επιμείνουμε σε αυτή τη θέση και την εξηγήσουμε, τότε μόνο μπορούμε να ε, στριμώξουμε κάπως το Συμβούλιο. Αν πούμε ναι, θα πρέπει να δεχτούμε γιατί πρέπει να καταλήξουμε κάπου, τότε θα βγούμε σίγουρα χαμένοι. Ελπίζω λοιπόν η διαπραγματευτική μας ομάδα να είναι σαφής, σαφής και κατηγορηματική και ο πρόεδρός μας να το πει και να στείλουμε τις, α, ε, ε, τις με web stream ή με το διαδίκτυο, το βίντεο από τη συζήτηση αυτή στο Συμβούλιο, γιατί φαίνεται δεν μπορεί να πάρει το αεροπλάνο από την Αθήνα για να έρθει να την παρακολουθήσει και να τη στείλουμε στι 28 κυβερνήσει και στη γερμανική κυβέρνηση τι ηχογραφήσει, να ακούσουν τι είπε το Κοινοβούλιο. Και ελπίζω να είμαστε συνεπείς και με την ψηφοφορία αργότερα. Δεν υπάρχει λύση που να περνάει από τη διακυβερνητική μέθοδο, γιατί η διακυβερνητική μέθοδος προστατεύει ε, τους, ε, δεν προστατεύει τους ε, φορολογούμενους αλλά τις ιδιωτικές τράπεζες και αυτό θα πρέπει να τονίσουμε στην προεκλογική μας εκστρατεία. Εκ μέρου των μεταρρυθμιστών συντηρητικών, ο κύριο Κάλαναν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσ... Εγώ προσπαθώ συνήθω να είμαι αισιόδοξο για αυτά τα ζητήματα. Κάποια μέρα πιστεύω ότι ακόμα ο κύριο Πον Μπέντι θα πει κάτι λογικό. Πριν από ένα χρόνο ακόμα και εγώ ήμουν σκεπτικιστής κατά πόσο θα κατέληγε το Συμβούλιο σε κάποια συμφωνία για τα θέματα στην τελευταία φάση της Τραπεζικής Ένωσης. Διότι εσείς είμαστε ρεαλιστές περί αυτού. Εδώ μιλάμε για πολύ σημαντική αλλαγή όσον αφορά την κυριαρχία στην Ευρωζώνη και μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλα ποσά χρηματικά. Ε, Έμαστε εν ώψη συμφωνία που θα δώσει απαιτούμενη ασφάλεια στι τράπεζε τη Ευρωζώνη. Σίγουρα αυτό είναι προ όφελο των πάντων. Ακόμα και αν δεν συμμετέχει η χώρα μου, πιστεύω ότι είναι προ δικό μα όφελο επίση αυτό να γίνει. Επίση, είναι προ όφελο των πάντων να σταματήσει η πρακτική που ακολουθούσαμε. Δηλαδή, οι τράπεζε κάνουν τα κέρδη, όμω αν καταρρεύσουν, τελικά πρέπει να πληρώνουν οι φορολογούμενοι. Εγώ δεν συμφωνώ με πολλέ από τι απόψει από αυτού. Η ομάδα μου δεν είναι αντίθετη με τα περισσότερα στοιχεία του κειμένου της Οικονομικής Επιτροπής, όμως έχουμε κάποιε σοβαρέ ανησυχίες όσον αφορά τη θέση του Κοινοβουλίου. Καταρχάς πιστεύω ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι χώρες εκείνες που είναι εκτός της Ευρωζώνης που έχουν πολλέ θηγατρικέ ε, στην Ευρωζώνη, όπω είναι η Τσεχική Δημοκρατία και η Σουηδία, να εμπλέκονται πλήρω στι αποφάσει που θα επηρεάσουν τα συμφέροντά του. Δεύτερον, πιστεύω ότι θα πρέπει να προστατεύσουμε ε, τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ενώση, να μην πρέπει να σώζει τράπεζε σε ένα νόμισμα που πολλές χώρες δεν θέλουν να χρησιμοποιήσουν. Αυτές είναι οι κόκκινες γραμμές και οι προτάσεις του Κοινοβουλίου έχουν αυτή τη στιγμή δεν εγγυώνται κάλυψη αυτών των ανησυχιών. Συμφωνώ με την ανάγκη όμω περί σαφηνία σχετικά με τη λήψη αποφάσεων. Ποιο θα αποφασίζει όταν θα χρεοκοπεί μια τράπεζα Ευρωζώνη. Και συμφωνώ οι ανησυχίε που ότι μερικέ μεγάλε χώρε θα μπορούν να ελέγχουν το πώ λειτουργεί αυτό ο μηχανισμό. Θα πρέπει όμω να είμαστε προσεκτικοί, να μην πάμε προ την αντίθετη κατεύθυνση και να δημιουργήσουμε τόσο άκαμπτη δομή που τελικά δεν θα μπορεί να τα αποκρίνεται ω ενδείκνυται στη όταν αποτυχάνουν οι τράπεζε, όταν καταραίουν οι τράπεζε οποτεδήποτε και οπουδήποτε. Άρα χρειάζονται βελτιώσει οι θέσει και του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου μέχρι ότου να βρούμε μια λύση η οποία να ταιριάζει και στι βόρειε και στι νότιε χώρε και στις χώρες Ευρωζώνης και στις χώρες που είναι εκτός Ευρωζώνης. Για κάποιους σήμερα η σημερινή συζήτηση και ψηφοφορία δεν είναι κάτι που αφορά εξέβρεση λύσης και να προχωρήσουμε, αλλά αφορά συσχετισμό δυνάμεων μεταξύ των θεσμικών οργάνων δυστυχώ. Και ο κ. Βεχόφστα που ίδιο είπε ότι κάποια αλλαγή πρέπει να αντιγράψουν οι ΗΠΑ των Αμερική. σω να το κάνουμε και αυτό και σε άλλου τομεί τη πολιτική. Η ομάδα μου δεν είναι απόλυτα ικανοποιημένη ούτε με τη θέση του Συμβουλίου ούτε με του Κοινοβουλίου. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να σεβόμαστε του κανόνε τη αγορά, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να σεβόμαστε του κανόνε περικατικών ενισχύσεων, όμω προσπαθήσαμε προσεγγίσουμε αυτά τα θέματα εξετάζοντας τη γενικότερη εικόνα που θα πρέπει να ξεπερνά τους μικροτσακωμούς, τους θεσμικούς, στους οποίους θέλουν να συμμετέχουν μερικοί. Σύμφωνα με τη συνθήκη της Αβώνας, αυτό το κοινοβούλιο έχει σημαντικές εξουσίες. Ας προσπαθήσουμε να τις ασκήσουμε αυτές τις εξουσίες με ευθύνη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Κάλλοναν. Τώρα εκ μέρους της Ελληνοτικής Αριστεράς, κυρία Τσίμερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο μηχανισμός εξυγίανσης για τις τράπεζες αποτελεί ουσιώδες τμήμα της Τραπεζικής Ένωσης. Άρα θα πρέπει και να φροντίζει ώστε να περιορίζονται οι υπερβολικές ε, συνέπειες που προκύπτουν από τη δυσλειτουργία τραπεζικού τομέα. Ωστόσο, εάν κοιτάξουμε τι προτάσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα και τα επιχειρήματα βέβαια από πλευρά του Συμβουλίου, αλλά και τη συζήτηση εδώ στο Κοινοβούλιο, μπορεί να έχουμε διατυπώσει μεγάλες, να έχουμε κάνει μεγάλες εξαγγελίες, μεγάλα λόγια, αλλά εν τέλει διαπιστώνουμε ότι όδινε είναι Και έτσι Κύριε Πρόεδρε, θα πρέπει πιστεύω εσείς να απευθυνθείτε στο Συμβούλιο, το οποίο λάμπει δια της απουσίας του σήμερα και να εξηγήσετε μέσω της ελληνικής προεδρίας ποια είναι ξεκάθαρα η θέση μας. Δεν νομίζω ότι καλύπτεται αυτή η απουσία από την παρουσία της Επιτροπής εδώ. Διότι οι επικρίσεις δεν απευθύνονται στην Επιτροπή. Η ομάδα μου, παραδείγματι, δεν είναι πεπισμένη ότι η απάντηση που λάβαμε από τον κύριο Μπαρόσο επί της δικής σας επιστολής αρκεί ως βάση. Γι' αυτό εγώ θα ήθελα μια σαφή τοποθέτηση και από την Επιτροπή για το ποιες είναι της θέση στην κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι διαπραγματεύσει τώρα και θα πρέπει να μας πει η Επιτροπή ξεκάθαρα τι πιστεύει και πώς μπορεί να επιτελέψει ουσιαστικά το ρόλο της ως θεματοφύλακα των συνθήκων. Αλλά για την κατάσταση των διαπραγματεύσεων. Έγινε χθε ε, ο τριμερής διάλογος, θα ακούσουμε φαντάζομαι και την αξιολόγηση, αλλά βλέπουμε ότι δεν υπάρχει καμία κινητικότητα από πλευρά του Συμβουλίου, ούτε ως προς τη διάσταση της διακυβερνητικής συμφωνίας, ούτε ως προς τη διάσταση που αφορά τη διαδικασία για τη λήψη αποφάσεων για την περίπτωση ε, εκαθάρισης. Εμείς λοιπόν θέλουμε να μείνει η νομική βάση στο άρθρο 114, την κοινοτική μέθοδο δηλαδή. Και πρέπει το Κοινοβούλιο να επισημάνει ξεκάθαρα ότι θα χρειαστεί να ληφθούν όλες οι σοβαρές αποφάσεις, όλες τις σημαντικές αποφάσεις με την συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί μπορεί να έχουμε και αλλού πιέσεις για τη διακυβερνητική μέθοδο. Θέλω λοιπόν να πω ξεκάθαρο ότι δεν είναι δεκτό την τελευταία απόφαση, την τελική απόφαση να τη λαμβάνει το Συμβούλιο, γιατί ξέρουμε πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα. Τα ισχυρότερα κράτη μέσα στο Συμβούλιο φροντίζουν να βρίσκουν λύσεις για το ίδια προς το συμφέρον των δικών τους τραπεζών, επιβάλλοντας τους κανόνες στους άλλους και έτσι εν τέλει εθνικοποιείται το ιδιωτικό χρέος των τραπεζών και επιβαρύνεται το κράτος μέλος, ο φορολογούμενος δηλαδή, να ε, επομιστεί το χρέος αυτό τα χρέη αυτά και ως εκ τούτου ενισχύονται οι ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών. Αυτό θέλω ιδιαίτερα να το υπογραμμίσω και υπογραμμίσω ότι δεν πρόκειται να δεχθούμε μια τέτοια πρόταση. Αλλά θα ήθελα και μια πιο βασική προσέγγιση, αυτό που είπα νωρίτερα ότι ε, όδιν εν όρος και έτε και μην. Όταν ε, κάνουμε τη συζήτηση με ορολογία too big to fail, ότι παρένει μεγάλο ε, οι τραπεζές για να αποτύχουν, ε, ουσιαστικά έχουμε χάσει την αντίληψη της υπόθεσης. Μιλούμε για περίπλοκους μηχανισμούς εξυγίανσης, αντί να πούμε ότι μια τράπεζα σε μικρότερες διαστάσεις μπορεί να κάνει τις ε, συναλλαγές για, την οποία, ε, για τις οποίες έχει σχεδιαστεί, για τις οποίες έχει συσταθεί και αν χρειαστεί να περάσει στη διαδικασία της εκαθάρισης. Αντί να μπαίνουμε σε διάφορους περίπλοκους μηχανισμούς. Μια άλλη παρατήρηση γιατί ακούσαμε από το Γερμανικό Υπουργείο των Οικονομικών ε, για μια έκθεση η οποία έλεγε ότι πραγματογνωμοσύνη είναι καλύτερα, ότι δεν αρκεί το άρθρο 114 ε, νομική βάση και ότι έπρεπε να υπάρχει και το 253. Δεν είναι καθόλου επαρκής αυτές οι επιχειρηματολογίες ε, του Γερμανικού Υπουργείου των Οικονομικών. Δεν εξηγείται πουθενά γιατί θα πρέπει να αποκλίνουμε από την αρχή την, ε, την, κοινοτική, ε, την κοινοτική μεθόδου με το άρθρο 114 και θα έλεγα ότι καλό θα ήταν στην γερμανική κυβέρνηση να μιλάει όχι μόνο το συντηρητικό σκέλος, αλλά και οι σοδημοκράτες πιο δυνατά, οι οποίοι πάντοτε δηλώνουν ότι, τουλάχιστον ιδιαίτερα τις τελευταίες εβδομάδες, ότι δεν πρόκειται να δεχθούν να συμπράξουν σε αυτή τη γερμανική κυβέρνηση, στο γερμανικό κυβερνητικό συνασπισμό, όταν επιβάλλει τη συντηρητική έποψη των ε, χριστιανοδημοκρατών μόνο σε ολόκληρο το Συμβούλιο. Ελπίζω λοιπόν στους σοδημοκράτες να επιδείξουν ε, την υπευθυνότητα που οφείλουν. Ο Πρόεδρος, παρακαλώ να ολοκληρώνεται. Και νομίζω ότι πρέπει να μην δεχθούμε να τεθούμε σε καθεστώ πίεση χρόνου, γιατί δεν έχουμε προξενήσει εμείς αυτή την καθυστέρηση, το Κοινοβούλιο δηλαδή. Την καθυστέρηση την χρεώνεται ολόκληρο το Συμβούλιο και αν πρόκειται να κλείσει η θητεία του Κοινοβουλίου χωρίς απόφαση, ε, κλείσει χωρί απόφαση και χωρίς καμία διαπραγμάτευση. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα εκ των ε, Ελευθέρων Δημοκρατών, ο κύριος Στέργο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θεωρώ ότι το πρώτο βήμα της Τραπεζικής Ένωσης ήταν καλό και καινοτόμο. Στο δεύτερο όμως βήμα, στο δεύτερο στάδιο, έχω πολύ σοβαρές επιφυλάξεις. Οι οικονομολόγοι πιθανολογούν ότι με ένα ταμείο με τόσους λίγους πόρους ε, το όλο σύστημα δεν θα είναι αποτελεσματικό. Και με απασχολεί το θέμα της κοινή ευθύνης του μηχανισμού εξυγένσης που εμπλέκει και τις κυβερνήσεις. Είναι σαφές ότι τα κράτη-μέλη θέλουν να αποφύγουν ένα σύστημα κοινή ανάληψης ευθυνών για τις τράπεζες ή τα χρηματοπιστωτικά του ιδρύματα πρέπει να πούμε στους πολίτες ε, ότι με το σύστημα αυτό θα εξοικονομήσουμε δαπάνες. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Αν θεσπιστεί το Ταμείο των Τραπεζών, το κόστος θα μεταφερθεί από τις τράπεζες, ε, θα, το μετακυλήσουν οι τράπεζες ε, στα τέλη και στις προμήθειες που εισπράττουν. Οπότε ουσιαστικά στους πολίτες. Ούτε είναι σίγουρο ότι θα αποτρέψουμε μελλοντικές κρίσεις χωρίς τη συμμετοχή των φορολογουμένων. Οι φορολογούμενοι πάντα πληρώνουν, είτε πρόκειται για κρίση είτε όχι. Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα. Και αυτό με προβληματίζει γιατί όποιο βιάζεται σκοντάφτει. Αν θέλουμε ένα ταμείο που θα ιδρυθεί και θα ασχίσει να λειτουργεί το συντομότερο δυνατό, αυτό δεν θα πρέπει να αποβεί βάρος των διαπραγματεύσεων. Θα πρέπει να προβλέψουμε χρόνο για τη σωστή θέσπιση και λειτουργία του Ταμείου. Και δεν είναι υπερβολικό διάστημα ή δεκαετία. Άλλωστε, η χρεοκοπία μια τράπεζα είναι μια περίπλοκη διαδικασία σε κάθε χώρα. Στη δική μου πατρίδα, τη Φιλανδία, έχουμε τρει μεγάλε τράπεζε. Οι δύο δραστηριοποιούνται και σε άλλε σκανδιναβικέ χώρε. Η Σουηδία όμω και η Δανία δεν συμμετέχουν στον μηχανισμό αυτό. Τι θα συμβεί αν αυτέ ε, οι σκανδιναβικέ τράπεζε ε, αντιμετωπίσουν προβλήματα φερεγγιότητας προς το παρόν είναι μια χαρά. Αλλά τι θα γίνει αν αντιμετωπίσουν προβλήματα στο μέλλον. Πώς θα έχει η κατάσταση στις διάφορες χώρες. Πολύ φοβόμαστε ότι εμείς θα πληρώσουμε την ύφη. Και πάνω απ' όλα με φοβίζει αυτή η επίσπευση της διαδικασίας. Ε, δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι ο μηχανισμός αυτός στόχο έχει να αποτρέψει τις μελλοντικές κρίσεις και όχι να αντιμετωπίσει την τρέχουσα. Άλλωστε, τα τοξικά δάνεια και οι τοξικοί ισολογισμοί δεν εντάσσονται στο μηχανισμό αυτό. Άλλωστε απέτυχαν και τα τεστ ε, αντοχής για τις τράπεζες. Ε, η διαμόρφωση μιας ε, σωστής τραπεζικής ένωσης δεν θα γίνει άρον-άρον με την αποφυγή πολιτικής ευθύνης. Θα γίνει με σωστή διαπραγμάτευση. Ευχαριστώ πολύ, κύριο Στόιανοφ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στη δουλειά που έχω κάνει εδώ σε αυτή τη θητεία, πάντοτε αγωνίζομαι να προστατέψω τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτών των πολιτών που μας βλέπουν εδώ από τα θεωρία. Που κάθε μέρα εργάζονται για να προκόψουν. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όπως κάθε άλλος πολίτης, θέλει να έχει ασφαλείς καταθέσεις, θέλει να μην πληρώνει διπλά τα λάθη των καρχαριών αυτών των αχόρταγων τραπεζιτών και έχει έρθει πια η στιγμή πιστεύω να λάβουμε μια στεναρή απόφαση να υπενθυμίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μία κυρίαρχη ένωση κρατών, όχι μια ένωση 28 αυτόνομων επαρχιών και υποστηρίζω τον κύριο Σφόμποντα που λέει ότι δεν μπορούμε να αποκλείσουμε κάποια κράτη για ορισμένους λόγους αν υπάρχει ένας ενιαίος ρυθμιστικός μηχανισμός, ένας ενιαίος ε, μηχανισμός που πρέπει να εφαρμόστε με τον ίδιο όρο σε όλους, με τους ίδιους όρους σε όλους, αλλά δεν έχει αρμοδιότητες η Ευρωπαϊκή Ένωση να δράσει εδώ. Και αν ένα από τα κράτη-μέλη και μάλιστα το μεγαλύτερο. Εκεί δηλαδή στο οποίο εδρεύει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εάν αυτό το μεγάλο κράτος θεωρεί ότι το ενοχλεί κάτι σε σχέση με αυτές τις προτάσεις, τότε πρέπει όλοι μας να διερωτηθούμε τι πάει στραβά. Κατά τα άλλα υποστήριζω τους ομιλητές και συναδέλφους και η δουλειά μου όλη δείχνει πως έχω από την αρχή στηρίξει την έκθεση αυτή. Ωστόσο, αν θέλουμε το σύστημα αυτό να φέρει αποτελέσματα για τον κάθε ένα, θα πρέπει να γίνει μεταρρύθμιση των συνθήκων. Πρέπει να τροποποιηθούν οι συνθήκες και όλα τα κρατη μπορούν πια, εφόσον οι κυρίαρχοι λαοί εγκρίνουν τις συνθήκες, θα πρέπει να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο κάποιου τύπου πονδιοποίηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Σούπερ Μάριο, ο Ντράγκη δηλαδή, έχουν πια ξεφύγει. Γιατί θα θυμίσω ότι δεν βρισκόμαστε σε κανένα ηλεκτρονικό παιχνίδι εδώ πέρα. Δεν προσπαθούμε να πυροβολήσουμε πάνω σε ψηφιακά μανιτάρια. Έχουμε να κάνουμε δουλειά για μια ουσιαστική κυρίαρχη ένωση. Ευχαριστώ κυρία Μπόλς. Ευχαριστώ. Ακούσαμε από τους προέδρους της ομάδας που ενισχύαν τη θέση της ε, Επιτροπής μου και αυτά που είπαμε στη συζήτηση περισμένης εβδομάδας, στους τριμερείς διαλόγους, στήριξα και θα υποστηρίξω ότι όλα τα θέματα είναι επιτάπητος όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις. Έγιναν τρεις τριμερείς διάλογοι όπου η ελληνική προεδρία δεν είχε διαπραγματευτική εντολή πέραν από αυτή τη θέση του Συμβουλίου. Και υπάρχουν όρια όσον αφορά το για πόσο μπορούμε να εξηγούμε ο ένας τη θέση του άλλου. Και έτσι χάνουμε χρόνο. Εγώ ανέλαβα πρωτοβουλία δική μου και έδωσα ιδέε πέραν από αυτέ τι θέση του Κοινοβουλίου. Προσπάθησα να είμαι τολμηρή και να προσπαθήσω και βοήθησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά χρειάζονται και δύο πλευρέ για να κινηθεί το θέμα. Δεν μπορώ να οδηγώ σε μονόδρομο του συναδέλφους και δεν έχω όρεξη ούτε πρόθεση να κάνω κάτι τέτοιο. Λοιπόν, το Συμβούλιο θα πρέπει να κινηθεί και να χρησιμοποιήσει και αυτό τη φαντασία του και να είναι περισσότερο ευρωπαϊκό. Και να είμαστε σαφές ότι μικρά σταδιακά βήματα δεν αρκούν. Κάποιοι υπουργοί είπαν ότι δεν υπάρχει ευελιξία. Δεν λειτουργεί έτσι το σύστημα. Υπάρχουν ωφέλη και θετικά στοιχεία στις προτάσεις και στι θέσεις του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου και στις δύο θέσεις. Και αν θέλουμε να έχουμε αυτό τον νέο μηχανισμό εξυγίανσης, δέχομαι ότι θα πρέπει να έχουμε το καλύτερο και από τι δύο θέσεις. Δεν είναι το καλύτερο ή το χειρότερο από τη μία πλευρά και μόνο. Συναπόφαση σημαίνει ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε το βέλτιστο μείγμα και από τι δύο θέσεις. Μπορούμε να δείξουμε σήμερα ότι μπορούμε να ψηφίσουμε μόνο τη θέση τη μία πλευρά. Μπορούμε να επανέλθουμε και να ψηφίσουμε δίκαιο συμβιβασμό. Αλλά δεν θα επανέλθουμε να ψηφίσουμε τη θέση του Συμβουλίου ή σχεδόν ταυτόσιμη εκδοχή αυτής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Μπόλς και τώρα εκ μέρου της κυρίας Φεραίρα η συγγήτριας ο κύριος Σάντσος Πρεσέδου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εκ μέρου τη κυριας φεραιρα η συγγητρια ο κύριο Σάντσο πρεσεδου ευχαριστω κυριε προεδρε εκ μερου της συγγητριας Ελίσσα φεραιρα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφου ε, για τη συζήτηση που έκαναν. Κύριε Σάντσες, με συγχωρείτε, θα σας διακόψω για ένα λεπτό. Κύριε Λάγκεν, το αντελήφθην και εγώ σας ευχαριστώ για την ευγενική υπόδειξη. Η γερμανική καμπίνα σήμερα φαίνεται ότι αντιμετωπίζει τεχνικά προβλήματα Ωραία. Ακούμε και πάλι τα γερμανικά. Περάστε κύριε Σάντσος, Πρεσέντο. Συνεχίζω λοιπόν κύριε Πρόεδρε. Είπα στην αρχή ότι ευχαριστώ τους συναδέλφους για το ύφος και το περιεχόμενο της συζήτησης που έγινε επευκαιρία της παρουσίασης ε, της θέσης της, πολιτικής οικονομικών, της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων και ευχαριστώ και τους συναδέλφους ε, που έλαβαν το λόγο εκ μέρους των πολιτικών ομάδων. Ναι, κύριε Σάρτσος πιστεύω σας διακόπτω και πάλι. Λυπούμε, λυπούμε πάρα πολύ. Η γερμανική καμπίνα μου λέει ότι κάποιος τους παίρνει το μικρόφωνο. Ποιος κλέβει το μικρόφωνο των Γερμανών, πείτε μου ποιοι είναι αυτοί οι κακοποιοί. Οι Βρετανοί. Λοιπόν, το United Kingdom παρακαλώ να μείνει στην καμπίνα του και να αφήσει και τη γερμανική καμπίνα να κάνει τη δουλειά τη. Κύριε Σάντσε Πρεσέντο, σα ζητώ και πάλι συγγνώμη για τη διακοπή. Φυσικά. Όλοι μας ενδιαφερόμαστε για την εύρυθμη λειτουργία της, ε, του γερμανικού καναλιού και της γερμανικής καμπίνας. Όπως ακούσαμε, δεν είχαμε κανένα αποτέλεσμα από τους τριμερείς διαλόγους μέχρι τώρα. Οπότε θα πρέπει να γίνουν κάποιες ψηφοφορίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να ψηφίσουμε με τρόπο ώστε να επομιστούμε τις ευθύνες μας ως συνομοθέτες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης, να φροντίσουμε η νομοθετική ρυθμίση να έχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και μάλιστα να φαίνεται αυτό με σαφή και κατηγορηματικό τρόπο. Η Τραπεζική Ένωση θα πρέπει να είναι τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα ενωσιακό σχέδιο. Χρειαζόμαστε ένα ενιαίο μηχανισμό που θα επεμβαίνει άμεσα και χρειαζόμαστε και ένα ενιαίο ταμείο που θα λειτουργεί από την πρώτη στιγμή και θα είναι εφοδιασμένο και με ένα προπολογισμό. Επίση, θέλουμε να απευθύνουμε έκκληση προ το Συμβούλιο να δώσει διαπραγματευτική εντολή στην Ελληνική Προεδρία. Γιατί η βούληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι να καταλήξουμε σε συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση, αλλά μια συμφωνία που θα είναι ουσιαστική αλλά και φιλόδοξη. Γι' αυτό και θεωρώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει αυτή τη στιγμή να λάβει το λόγο και να απευθύνει μια έκκληση στο Συμβούλιο. Και περιμένουμε την απάντηση και την αντίδραση του Συμβουλίου. Ευχαριστώ εκ νέου Επιτροπή ο κύριος Μπαρνί. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και καλημέρα σε όλους τους παρισταμένους κυρίες και κύριοι βουλευτές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που με καλέσατε να μιλήσω και πάλι αυτήν την εβδομάδα για το σημαντικό αυτό θέμα και ιδιαίτερα στο πλαίσιο της Τραπεζικής Ένωσης, στο σημαντικό αυτό πυλώνα, αφού χτίσαμε τον πρώτο πυλώνα που είναι η εποπτεία των, τραπεζικών της, των τραπεζών της Ένωσης και εκείνων όσα θα ήθελαν να ενταχθούν στην Τραπεζική Ένωση χωρίς να έχουν ή πριν να ενταχθούν στο ευρώ. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι όπως και στο περιβάλλον η πρόληψη κοστίζει λιγότερο από την αποκατάσταση. Η εποπτεία σημαίνει πρόληψη. Όταν όμως πρέπει παρόλα αυτά να αποκαταστήσουμε μια ζημιά, πάντα είναι καλύτερο να είμαστε προετοιμασμένοι για την επιδιόρθωση, την αποκατάσταση. Η προπαρασκευασμένη και οργανωμένη επιδιόρθωση κοστίζει λιγότερο από την άτακτη μη οργανωμένη που επιβαρύνει περισσότερο το φορολογούμενο. Και γι' αυτό θα ήθελα και να υπογραμμίσω από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή πω. Πιστεύουμε ακράδαντα πως ε, το θέμα το οποίο συζητούμε είναι κατεπήγον να προχωρήσει το ταχύτερο δυνατό. Τόσο η Επιτροπή όσο και το Κοινοβούλιο επιθυμούν μια καλή συμφωνία, μια συμφωνία αξιόπιστη για τη λειτουργία της, μια αξιοπιστή αξιόπιστη και για τους παράγοντες των χρηματοπιστωτικών αγορών που θα θεσπίσει ένα μηχανισμό ε, υγιή, στεναρό, αποτελεσματικό και που όταν χρειαστεί ομιγένετο θα οδηγεί σε μια τακτική διαδικασία καθάρισης των τραπεζών χωρίς να γίνεται ε, τακτικά και συστηματικά απομίζηση των ε, φορολογουμένων. Χωρίς να στάνε δηλαδή από τους φορολογούμενους να βάλουν το χέρι στην τσέπη όπως έλεγε ο κύριος Τέχτο νωρίτερα. Και υπενθυμίζω ότι το κείμενό σας και βέβαια ο τριμερής διάλογος με την κυρία ε, Sharon Μπόλ, την κυρία Βόρτμαν Κόλ, την κυρία Φόρτ, τον κύριο Σάντσες Πρεσέντο, την, ε, τον κύριο Γκίκολτ και το λέω κύριε Πρόεδρε εδώ γιατί ιδιαίτερα πρέπει να απευθύνω θερμούς χαιρετισμού και ευχές για ταχύτατη ανάρρωση προς την κυρία Φερέιρα που έχει κάνει τόσο πολύ καλή δουλειά οι ευχέ λοιπόν βγαίνουν και από τα τείχη του Κοινοβουλίου και πιο έξω και θέλουμε έναν ε, ανοιχτό μηχανισμό όπως είπε και ο κύριος Βενιζέλος νωρίτερα. Θέλουμε λοιπόν μία ε, ε, επανεξετάσαμε τεχνικά σημεία του κειμένου, ένα κείμενο πολύ περίπλοκο με σημαντικά διακυβεύματα και ως εκ τούτου απαιτείται συζήτηση επί της ουσίας. Υπενθυμίζω ότι μιλούμε για εκαθάριση τραπεζικών ιδρυμάτων που χρηματοδοτούν κατά 75% τα κράτη τις ε, περιφερειακές τοπικές ε, οργανώσεις, τους πολίτες, τις επιχειρήσεις των κρατών. Και άρα έχουν τεράστια συνέπεια τα προβλήματα που αυτές θα αντιμετωπίσουν ε, στην οικονομία και τη ζωή των πολιτών. Άρα λοιπόν πρέπει χωρίς να καθυστερούμε, όπω είπε η κυρία Βόρτμαν Κόλ, να αναλάβουμε δράση. Ο κύριο Φερχόφστατ δεν είναι εδώ τώρα. Μιλούσε ολότερα για τα διδάγματα από την κρίση. Σε περίοδο κρίση, και α είμαστε και έντιμοι, κυρίε και κύριοι βουλευτέ, με τη δουλειά που έχετε κάνει εσεί, που έχετε κάνει το Συμβούλιο και εγώ όσο μπορούσαμε τι ε, ομάδε όλε, έχουμε κάνει ό,τι μπορούσαμε για να αντλήσουμε και τα σωστά διδάγματα από την κρίση. Πάνω από 30 νομοθετήματα ε, εκπονήθηκαν και εγκρίθηκαν ως αποτέλεσμα και ως συνέπεια της κρίσης, όπως κάναν και οι Αμερικανοί από την άλλη μεριά του Ατλαντικού, προσπαθούμε και εμείς να προστατέψουμε τον καταθέτη, τον ε, πολίτη, τον φορολογούμενο. Δεν έχουμε τελειώσει αυτή τη δουλειά ακόμα. Έχει μείνει αυτός ο δεύτερος πυλώνας της Τραπεζικής Ένωσης και για την κυρία Τσίμερ, που δεν με παρακολουθεί, αλλά φαντάζομαι ότι θα ενημερωθεί από τα πρακτικά. Φίλεν Dank. Μόνο και μόνο επειδή και εγώ σας άκουσα και θα ήθελα να σας πω ότι ε, θα ήθελα να δώσετε προσοχή στο τελευταίο κείμενο που παρουσίασα την προηγούμενη εβδομάδα στην Επιτροπή για τη διαρθρωτική μεταρρύθμιση των 30 μεγαλύτερων τραπεζών. Γιατί ακριβώ αυτό το θέμα θέλουμε να αντιμετωπίσουμε, το πρόβλημα των μεγάλων τραπεζών και να τι ενθαρρύνουμε να κάνουν τη δουλειά τους, όπως είπατε και εσείς κυρία Τσίμερ, να ε, κάνουν τη δουλειά τους δηλαδή να δανείζουν σε επιχειρήσεις, να, δίνουν, να δανείζουν στον καταναλωτή και όχι να κερδοσκοπούν. Και πρέπει να είμαστε έντιμοι, πολλή δουλειά ακόμα μένει να γίνει για να καταλήξουμε σε συμφωνία. Καταρχάς έχουμε το κεντρικό και πολύ λεπτό αυτό ζήτημα και κρίσιμο ζήτημα για το Κοινοβούλιο της διακρατικής, της διακυβερνητικής συμφωνίας ε, που ζητά το Συμβούλιο σας είπα την τρίτη ποια ήταν η θέση της Επιτροπής. Είμαστε πεπισμένοι, κύριε και κύριοι βουλευτέ, ότι το άρθρο 114 είναι η σωστή νομική βάση και κύριε Στογιάννοφ έχουμε βάση για να δράσουμε. Το είπα και το επαναλαμβάνω, το άρθρο 114 για την ε, ίδρυση του Ταμείου Εκαθάρισης Εξυγίανσης. Θα ήθελα επίση να υπογραμμίσω και να προσθέσω ότι η, πρόσβα, η, προσφυγή σε μια τέτοια συμφωνία δεν είναι αντίθετη με την συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν αφορά την ε, μεταφορά και την αμοιβαία χρήση των κονδύλιων. Και κυρία Τσίμερ, μια και εσείς με ρωτήσατε, ο πρόεδρος ε, Μπαρόσο απάντησε στον ε, πρόεδρο Σούλτς και είμαι και εγώ στη θέση όπω και χτες με τον τριμερή διάλογο για να διευκρινίσουμε τις διαφορετικές τοποθετήσεις και να δώσουμε απαντήσεις στα νομικά ακόμη ζητήματα. γι' αυτό και να είμαστε σαφείς ότι αν αποφασίσει τελικά το Κοινοβούλιο να επιδείξει ε, πνεύμα διαπραγμάτευση, συμβιβασμού στο τόσο σημαντικό αυτό θέμα, το Συμβουλίο και ελπίζω να μας παρακολουθεί, θα δείξει, θα επιδείξει την εκτίμησή του και στο μέτρο που χρειάζεται θα καταλήξει στα σωστά συμπεράσματα για κάθε άλλη πτυχή της διαπραγμάτευσης. Εν προκειμένου υπάρχουν σημεία του μηχανισμού εξυγίανσης που θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης και αποφάσεων αλλά και όλα τα θέματα, όπως είπε η κυρία Σάρον Μπόλς νωρίτερα, ε, που χρήζουν ακόμη συστήσεως. Χρηματοδότηση, διακυβέρνηση, δημοκρατική λογοδοσία του Συμβουλίου, του Συμβουλίου Εξυγένσης, όλα αυτά τα θέματα που σας ανέφερα νωρίτερα. Και υπενθυμίσω τις κύριες πτυχές. Πρώτον, θα μπορούσαμε να αναλογιστούμε το ενδεχόμενο για μια επιτάχυνση της ε, ε, αμοιβαία διάθεση των ποσών ε, για να φτάσουμε το ταχύτερο δυνατό σε ένα κοινό ταμείο και επίσης όπως είπε και η κυρία Βόρτσμαν ένα ταμείο κοινό από την πρώτη ημέρα και έτσι θα μπορούσαμε να απηχήσουμε και τις ιδέες του κύριου Φερχόφστατ για την ε, πρόβλεψη μιας περιορισμένης διάρκειας στη διακυβερνητική μέθοδο. Επίσης θα μπορούσαμε να αναφερθούμε στα backstops τους μηχανισμούς προστασίας. ακόμα και με αυτή τη διαδικασία της διάθεσης των κονδυλίων. Επίσης θα πρέπει να προβλέψουμε, θα πρέπει, μπορούσαμε να προβλέψουμε μηχανισμό που να επιτρέπει ταχύες και αποτελεσματικές αποφάσεις με ασφάλεια δικαίου, μια πραγματική δηλαδή ε, αποτελεσματικότητα στην, ε, στην απόφαση και τη δράση. Και κύριε Κάλλαναν, σ' άκουσα, άκουσα με προσοχή νωρίτερα και έχετε δίκιο. Πρέπει να είναι αποτελεσματικό αυτό ο μηχανισμό, να μπορεί να προβλέψει καταστάσει, να προλάβει καταστάσει και να αποτρέψει μια μεταγενέστερη κρίση, όχι μόνο να αποκαταστήσει αυτήν που ήδη έχει ξεκινήσει. Και επίσης θα πρέπει να ενισχυθεί η ε, δημοκρατική νομοποίηση του μηχανισμού που σκοπεύουμε να ιδρύσουμε και αυτό μπορούμε να το πράξουμε εμπνεόμενοι από τον εποπτικό μηχανισμό. Εν τέλει κυρίες και κύριοι και συντομία έχουν κατατεθεί όλες οι προτάσεις προ διαπραγμάτευση. Υπάρχουν φωνέ που μιλούν για συμβασμού. Πρέπει πια να, να προχωρήσουμε αποφασιστικά γιατί είναι περιορισμένο ο χρόνος. Ε, ξέρω ότι είναι διατεθειμένο το Κοινοβούλιο να προχωρήσει σε μια φιλόδοξη ε, λύση με έναν ε, στεναρό γερό μηχανισμό για τον καταθέτη, για τον φορολογούμενο, για όλη, όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και ως ε, Επίτροπο Αρμόδιο για την Εσωτερική Αγορά, θέλω ιδιαίτερα να επισημάνω ότι έχει σημασία η συνοχή και η λειτουργία τη εσωτερική αγορά. Υπάρχουν κράτη τα οποία δεν εντάχουν ενταχθεί ακόμη στο νέο νόμισμα και η σταθερότητα του ευρώ έχει εξίσου πολύ μεγάλη σημασία για όλου. Οι ίδιοι κανόνε λοιπόν θα πρέπει να ισχύουν για όλου, όπω και οι ε, κανόνε για τι κρατικέ ενισχύσει, για να διαφυλαχθεί η ενότητα και η συνάφεια, η συνοχή τη αγορά. Τη ενιαία αγορά. Πρέπει με, αυτούς, με αυτές αρχές να προχωρήσουμε, όπως είπε και ο κύριο Σφόποτα, όπω είπε και ο κύριος Φερχόφστατ επίση. Πρέπει να δοθεί μια νέα εντολή για το Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ. Αυτή την έκκληση απευθύνατε κι εσεί, αυτή την έκκληση μεταφέρω κι εγώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που πλευρά τη είναι διατεθειμένη να διαδραματίσει το ρόλο τη, θα συνεχίσει να τον διαδραματίζει. Ε, κινητοποιούμεθα, αναλαμβάνουμε δράση και έτσι μπορούμε να οικοδομήσουμε κυρίε και κύριοι βουλευτέ έναν αυθεντικά ευρωπαϊκό μηχανισμό, όπως είπε ο κύριος Κονπεντήτ, όπως είπατε και εσείς, ε, Πρόεδρος Φόμποντα, ένα μηχανισμό ο οποίος δεν θα υποκύπτει σε συμφερόντα και ε, ε, ε θέση ισχύω κάποιων κρατών. Πάντως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό θα αγωνιστεί. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ για τις δηλώσεις των ομάδων. Συμφωνούμε, φαντάζομαι, ότι η Τραπεζική Ένωση είναι ένα από τα σημαντικότερα, αν όχι το πιο σημαντικό, ε, εγχείρημα της τρέχουσας θητείας και η ολοκλήρωσή του με ένα μηχανισμό εξυγίανσης θα το καταστήσει ένα ιδιαίτερο εγχείρημα για την σταθερότητα όχι μόνο στην Ευρωζώνη αλλά ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κατάσταση λοιπόν είναι η εξής. Η Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το Δεκέμβριο προσδιορίσε τη θέση της με ψηφοφορία. Το Συμβούλιο όρισε τις δικές του θέσεις την επόμενη ημέρα. Και τώρα μεταξύ των δύο συνομοθετών πρέπει να ξεβρεθεί συμφωνία, μια λογική συμβαστική λύση που να εξασφαλίζει πλειοψηφία, Από τα όσα είπατε σήμερα ως πρόεδροι ε, ομάδων και της Επιτροπής των Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων. Βλέπω ότι θέλετε ιδιαίτερα να παραμείνει η διαδικασία στην, ε, στη δυνατότητα συμμετοχής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ιδιαίτερα θα ήθελα λοιπόν να υπογραμμίσω ότι αναφερθήκατε στην νομική ε, στην ε, νομιμοποίηση, δημοκρατική νομιμοποίηση και τη διαφάνεια, αλλά και στο γεγονό ότι δεν μπορεί να δεχθεί το Κοινοβούλιο να αποκλειστεί από την νομοθετική αυτή διαδικασία. Και με καλείται να αποστείλω επιστολή στο Συμβούλιο ε, με την οποία θα καλώ σε έκτακτη, θα ζητώ να διοργανωθεί μια έκτακτη συνεδρίαση του ΕΚΟΦΗΝ. Αυτό εκφράζουν με την ευρύτατη του πλειοψηφία οι ομάδε εδώ. Θα αποστείλω λοιπόν τη σχετική επιστολή στο Συμβούλιο και θα συμπληρώσω το κείμενο λέγοντα ότι ο κύριο Μπαρνιέ είναι έτοιμο να συμμετάσχει στι διαπραγματεύσει εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πιστεύω ότι το απόν Συμβούλιο μπορεί να ενημερωθεί με τον τρόπο αυτό, με την επιστολή μου δηλαδή, για αυτή την εξέλιξη. Herr Präsident, vielleicht kann mich Κύριε Πρόεδρε, ίσως μπορούσατε να μου εξηγήσετε τι είναι αυτή η παράξενη, παράδοξη, κομική διαδικασία για το θέμα αυτό, γιατί δεν καταλαβαίνω πολύ καλά. Έχει αποφασίσει η Επιτροπή να προχωρήσει σε τριμερή διάλογο και να μην γίνει ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο. Μετά ξεκινάμε τις συζητήσεις, πολύ ωραία μέχρι εκεί. Και τώρα σε αυτή τη θητεία δύο φορές συζητούμε εκτάκτως το ίδιο θέμα, σε δύο διαφορετικές μέρες. Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό. Και σήμερα λαμβάνεται απόφαση και επιπλέον αυτού θα αποστείλεται επιστολή, ενώ εκ παραλίλου συνεχίζει η φυσιολογική διαδικασία του διαλόγου, γιατί λοιπόν να διαλέγουμε ή τη μία ή την άλλη διαδικασία. Γιατί κάνουμε αυτό το, το υβρίδιο διαδικασία. Δεν καταλαβαίνω. Δεν το έχω ξαναδεί ποτέ. Υπάρχει κάποιο λόγο για τον οποίο το κάνουμε αυτό. Γιατί δεν ε, ακολουθούμε πιστά μία σαφή διαδικασία. Γιατί τα μπερδεύουμε. Γιατί αποκλίνουμε από αυτή την ξεκάθαρη διαδικασία και φοβάμαι ότι θα επαναληφθεί αυτό. Λοιπόν, εξηγήστε μου. Αυτό που είπατε αγαπητέ συνάδελφοι ότι ίσω να μην αντιλαμβάνεστε τα πράγματα το κρίνετε εσείς, δεν θα το κρίνω εγώ. Εν πάση περιπτώσει αυτή είναι η διαδικασία που ζητήθηκε, αυτή την οποία ακολουθώ εγώ, όπω τη ζήτησε η διάσκεψη των Προέδρων, η οποία μου είπε πριν από την Τετάρτη από τον τριμερή διάλογο να γίνει συνάντηση και αποφάσισε μετά τον τριμερή διάλογο, της Τετάρτης δηλαδή ε, χτες, τον χθεσινό, σήμερα το πρωί, να συναντηθεί με την διαπραγματευτική ομάδα, η διάσκεψη των Προέδρων, όπω και έγινε, και να γίνει ένας γύρος παρεμβάσεων από τους επικεφαλείς των πολιτικών ομάδων, όπως και έγινε, και με τα αποτελέσματα, για να ενημερωθούμε για τα αποτελέσματα του τριμερούς διαλόγου που έλαβε χώρα εχθέ, αυτό συνέβη σήμερα. Επίσης, η διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε και μάλιστα πριν από δύο εβδομάδες, 14 μέρες περίπου, είχε αποφασίσει η διάσκεψη των Προέδρων να υποβάλει στη ψηφοφορία τις τροπολογίες της ε, Οικονομικής και Νομισματικής Επιτροπής, χωρίς όμως τελική ψηφοφορία, με ε, σκεπτικό από πλευρά τη τύψη των Προέδρων ότι ήθελε να δείξει στο Συμβούλιο ποιε είναι οι θέσει ε, τη Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή και ότι τις στηρίζει τι θέσει αυτέ η Ολομέλεια και, και ω εκ τούτου με το σκεπτικό να ενισχύσει τη θέση των διαπραγματευτών εκ μέρους του Κοινοβουλίου στις ε, επαφές τους με το Συμβούλιο. Αυτό συμφωνήθηκε από τις περισσότερες ομάδες. Διαπιστώνω όμως ότι δεν είχατε από ό,τι φαίνεται ε, συνομιλήσει με τους διαπραγματευτές εκ μέρους του ΕΛΚ. Δεν ήσασταν ενήμερος. Όχι, εγώ σας ε, ενημέρωσα απλώς ότι εφαρμόζω όπως οφείλω τις αποφάσεις που έλεγε η διάσκεψη των Πρόεδρων. Κύριε Ρόιλ, κοιτάξτε, όχι, δεν ήταν καμία ανατροπή, ήταν απόφαση της διασκέψης των Προέδρων, την οποία ακολουθώ. Θέλει κάποιος άλλος το λόγο. κύριος Ο κύριος Σιμάνσκι. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ε, χθες πριν το τέλος ψηφοφορία ψηφοφορίας ε, της για την περιβαλλοντική και ενεργειακή πολιτική μέχρι το 2030 δεν με επέτρεψε ο Πρόεδρος να συμμετέχω στην τελική, στην τελική διαμόρφωση ε, και να έχω επιρροή στην τελική ψηφοφορία. Ε, το απόγευμα με ενημέρωσε το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι δεν τηρήθηκαν οι σωστές υποχρεώσεις για το θέμα αυτό. Θα ήθελα να ακούσω την επίσημη θέση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό, γιατί πραγματικά ε, ήταν τελείως αθέμητη αυτή η πρακτική και νομίζω ότι θα πρέπει να στυλιτευτεί και να τιμωρηθεί. Κύριε Σιμάνσκι, είναι αιτιολογημένη η παρέμβασή σας εχθές, πριν από την ψηφοφορία, είχατε ζητήσει το λόγο, γραπτά μάλιστα, από την προηγούμενη βραδιά. Και άρα έχετε δράσει σωστά. Οι υπηρεσίες της ε, Συνόδου ε, δεν μετέφεραν, έκαναν το λάθος να μην μεταφέρουν μέσα στο φάκελο της ε, Προεδρίας στον, στην αρμόδια αντιπρόεδρο την αίτησή σας και γι' αυτό παραλυφθήκατε. Το ανέφερα και σήμερα εγώ στη διάσκεψη των Προέδρων και ενημερώθηκαν. Ξέρετε, όταν δουλεύουν άνθρωποι συμβαίνει τέτοια λάθη. Οι υπηρεσίε λοιπόν τη Συνόδου, το γραφείο που οργανώνει τη Σύνοδο, έκανε το σχετικό λάθος και ζητεί συγγνώμη. Θα έπρεπε να έχετε λάβει όμω το λόγο, έχετε απόλυτα δίκιο, γιατί είχατε καταθέσει εγκαιρό στο αίτημα. Uh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το διαδικαστικό μου είναι το εξή. Η διάσκεψη των Προέδρων πήρε μια απόφαση περί αναβολής συζητήσεως σήμερα όσον αφορά τις καταστροφές που έχουν σημειωθεί στις δυτικές ακτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ενωμένο Βασίλειο, όλος ιδιαίτερος, σαν αποτέλεσμα των συνεχιζομένων καταιγίδων άνευ προηγουμένων και των πλημμυρών που έχουν επηρεάσει πάρα πολύ τι ζωέ των ανθρώπων. Θα έπρεπε τώρα να γίνει μια επίκαιρη συζήτηση για να δείξουμε μια αλληλεγγύη προ αυτού. Ήθελα να ξέρω γιατί αναβάλλεται αυτή η συζήτηση, εφόσον υπήρξε και μια κάποια παύση στη διαδικασία σήμερα. Μεταξύ 10.30 και 11 δεν έγινε κάποια προγραμματισμένη συζήτηση, υπήρχε χρόνο. Θα επαναπρογραμματιστεί για την επόμενη σύνοδο και θα εκφράσουμε αλληλεγγύη για τους πληγέντες ανθρώπους και να διαθέσουμε κάθε δυνατό μέσο για να του βοηθήσουμε αυτού του ανθρώπου. Το ανέφερε αυτό ο Ισπανό συνάδελφο εχθέ. Κύριε Κέλλη, και εδώ έχουμε να κάνουμε απόφαση τη σύψη των Πρόεδρων. Οι ομάδε δεν θέλησαν να μπει το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη για σήμερα. Αλλά, ανά πάσα στιγμή, μπορεί να επανέλθει στην ημερήσια διάταξη από ό,τι αντιλαμβάνομαι, πρόκειται να επιληφθεί και πάλι η αρμόδια καθήλυνη επιτροπή. Επομένω, κατά πάσα πιθανότητα θα το δούμε στην ημέρησια εντάταξη στην επόμενη σύνοδο. Κύριο Γκόλνιχ. Με συγχωρείτε κύριε Γκόλνιχ. Ένα λεπτό, με συγχωρείτε κύριε Γκόλνιχ. Στο ίδιο θέμα κύριε Σφόποντα, για την παρατήρηση του κύριου Κέλλη, παρακαλώ. Θέλω απλώς να πω στον κύριο Κέλλη ότι ήδη έχει προβλεφθεί έτοιμα για συμπερίληψη του θέματος στην προσεχή σύνοδο, γιατί υπάρχουν και άλλες περιοχές, Αυστρία, Ιταλία, που έχουν αντιμετωπίσει σοβαρέ χιονοπτώσει και μεγάλε πλημμύρε και έχουμε ζητήσει να προβλεφθεί στην μερίσια διάταξη τη προσεχή συνόδου. Προσεχού συνόδου, Άρα είμαι βέβαιο ότι θα υποστηριχθεί το αίτημα αυτό. Κύριε Γκολνίση, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομο. Είναι πολύ ευτυχέ το ότι έχετε στα καθήκοντά σας αναγνωρίσει, στα πέστη των καθηκόντων, αναγνωρίσατε το σφάλμα που έγινε βάση του κ. Σιμάνσκι. Επιτρέψτε μου όμως να σας πω ότι αυτό που αναμένεται από πλευράς κάποιων μελών του Κοινοβουλίου ε, δεν είναι δικαιολογίε τόσο πολύ. Ο κ. Σιμάνσκι ανακοίνωσε ότι ο συγητή συνέστη είναι καταψήφιση του κειμένου. Αυτό που είναι αρκετά σπάνιο. Και αυτό που θα, ε, θα γινόταν, εάν γινόταν η παρέμβασή του, θα είχε αποφασιστική σημασία για την ψηφοφορία. Οπότε, νο, θεμητά μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η ψηφοφορία ε, δεν έγινε σωστά, διότι δεν τηρήθη ο κανονισμός που έδινε το δικαίωμα λόγου στον εισηγητή. Και πιστεύω ψηφοφορία θα έπρεπε να επαναληφθεί για το λόγο αυτό. Ευχαριστώ. Yeah, Κύριε Το θέμα αυτό το συζητήσαμε. Το επαληθεύσαμε με πολύ μεγάλη προσοχή.